προεδρεύω τώρα. Αν είμαι ο παλιότερο ε, στην Επιτροπή αυτή, ο πιο ηλικιωμένο, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το οποίο οδήγησε στο να είμαι ε, ο προεδρεύων, αλλά είναι πράγματι μια μεγάλη τιμή, γιατί ήμουνα ακριβώ σε αυτή την αίθουσα πρόεδρο του ΕΛΚ για πάρα πολλά χρόνια και νιώθω μια ιδιαίτερη και βαθιά νοσταλγία που έχω αυτή την ευκαιρία να προεδρεύω και πάλι. Έχουμε όμω τώρα στην ημέρηση διάταξη. Έχετε σχόλια για την ημέρηση διάταξη. Όχι, δεν έχετε τότε εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Ερχόμαστε στην σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω απολύτω τίποτα εδώ. Δεν σταματάμε όμω εδώ. Περνάμε στην πρόταση για συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας για την απλούστευση της έκδοση προξενικών θεωρήσεων. Δεν έχουμε καθόλου τροπολογίε, έχουμε απλώ μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ παρακαλώ, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Νίλσεν. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Το θέμα που θέλω να εγείρω, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία για τη γνωμοδότηση αυτή να συζητήσουμε, θέλω να θέσω το εξή ερώτημα προς τον εισηγητή και προς την Επιτροπή μας. Όταν το Κοινοβούλιο συζήτησε τη συμφωνία αυτή για τη διευκόλυνση των προξενικών θεωρήσεων με τη Ρωσία, είχαμε ζητήσει αυτή η συμφωνία να μην εφαρμόζεται σε αυτούς που διαμένουν στις, στα εδάφη της Γεωργίας, της αυχαζίας και της Νοτίας Οσετίας που έχουν ρωσικά διαβατήρια. Θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν έχει σκεφτεί για την αντίστοιχη περίπτωση που ισχύει στην Αρμενία και εάν η συμφωνία αυτή διευκόλυνσης προξενικών θεωρήσεων θα περιλαμβάνει και τους κατοίκους του Άνω Καραμπάχ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Ο κύριος Πορέμπα, ο εισηγητής μας δεν είναι παρόν. Γι' αυτό ζητώ από την κυρία Νίλσεν να... να... ζητώ να, ο εισηγητής να δώσει μια γραπτή απάντηση στην κυρία Νίλσεν. Ερχόμαστε λοιπόν στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία όπως έλεγα ηλεκτρονικά. Πέρας. Παρακαλώ. Αρχίζουμε και πάλι την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Όλοι, όλες. Ο κύριος Πόσελ ψάχνει ακόμα την κάρτα του, αλλά κατά τα άλλα νομίζω οι υπόλοιποι έχουν ψηφίσει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. 28, 28 πράγματι. Με την κυρία Όμεν η οποία δεν είχε την κάρτα της. Ερχόμαστε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια. <clears throat> Πάλι δεν υπάρχει τροπολογία. Κύριε Λαντσπέργκης. Uh, uh, uh, for some information. is... Ζητώ μια πληροφορία. Έχει γίνει μια αντίστοιχη συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν ή όχι. Ή είναι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Πληροφορήστε με παρακαλώ. It's only Armenia at the moment. μόνο Αρμενία παρακαλώ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ήταν η ίδια διαδικασία αυτή που ίσχυσε για το Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ, λέει κυρία Γιάχτεμάκη. Εγώ είμαι η εισηγήτρια για το Αζερβαϊτζάν, για τη συμφωνία αυτή. Δυστυχώ όμως, Δυστυχώ, δεν, δεν έχω να σας πω κάτι για το θέμα αυτό. Δεν έχει προχωρήσει η απόφαση αυτή τη συμφωνία με την ταχύτητα που έχει συναυθεί η συμφωνία με την Αρμενία. Η ελπίδα μου είναι ότι ταχύτερα δυνατό θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε να επικυρώσουμε μια συμφωνία επανιστοχής με το Αζερμπαϊτζάν. Νομίζω ότι σας ικανοποιεί αυτό κύριε Λανσμπέργκης. Ναι, ναι, είναι σωστή η απάντηση, λέει ο κύριος Λαντσπέργης. Συνεχίζουμε, έχουμε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Κύριε Γκάλερ, θέλετε να ψηφίσετε. Ναι, ναι. Καθίστε λοιπόν. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Και η Ρία προστίθεται, 28 λοιπόν υπέρ, πάλι με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται να σας λέω κάθε φορά τα αποτελέσματα, τα βλέπετε. Στη συνέχεια. Διαφθορά στον δημόσιο και ειδικοτικό τομέα, επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες. Ε, τροπολογία 61, ψήφι υπέρ. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Για το δεύτερο έλεγχος, βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 61. Ευχαριστώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τρίτο τμήμα, πάλι ηλεκτρονικά, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 68 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72 υπέρ κατά. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσανε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεν ναι, εμπερδευτήκαμε ναι, λιγάκι, εν πάση έχει γίνει δεκτή. Συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 75 υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η παράγραφος 15 μάλλον η τροπολογία 96 τρία τμήματα πρώτο τμήμα δύο τμήματα δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές δεκτή 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ, επαναλαμβάνω. Κατά. Αποχές δεκτή. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι. Σύμφωνοι. Θέλετε έλεγχο. Ηλεκτρονικά. Συμβιβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. 104 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 20. Συμβαστική 20 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εντάξει, ήταν σαφές. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι 19, όχι δεν την ψηφίζουμε καλύπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23. 22 όχι. 22 εκπίπτει. 22 εκπίπτει. Πάμε στην 23. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 24 συμβατή με την 23. Ψηφίσουμε την 24. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε την 25 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πράγματι εγκρίνεται. Δεν ήταν φανερό από την αρχή. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε για την 29. Ναι, ναι. 29. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. <coughs> Με ισοψηφία. Καλά που ψηφίσαμε ηλεκτρονικά. 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και εδώ θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχιδε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά ηλεκτρονικά για τη 43 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρασε Ναι, ναι, πέρασε παρόλα αυτά. 15-14. 44 ναι, υπέρ. Κατά αποχές δεκτής. 45 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικά. 45 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ναι, ναι, εντάξει. 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά ηλεκτρονικά 47 άρχεται όλοι ψηφίσατε πέρας ισοψηφία απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ απορρίφθηκε θέλετε έλεγχο Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 58, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται, πράγματι. <coughs> Με υψοψηφία. 59, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή τέσσερα υπέρ κατά έλεγχος αρχίζει η ψηφοφορία για την τέσσερα. ψήφισατε όλοι πέρας δεκτή <laughs> όταν λέω αν έχει αν έχετε ψηφίσει όλοι και όλε θέλω να πω, αλλά δεν μπορώ να το λέω συνέχεια, μαλλιάζει η γλώσσα μου. 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά για την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε Πέρα. Πέρας. 15-15 απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ένα είναι γλωσσικού χαρακτήρα. Δεν την ψηφίζουμε. Γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Όχι. ΔΕΒΕ 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την ΔΕΒΕ 9. Ψηφίσατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. 15-15 απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕ 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ΔΕΒΕ 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΔΕΒΕ 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 28 υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές. Ταυμάσια. Συγχαρητήρια. Σαν τους παλιούς καλούς καιρούς που προέδρευα στη συνεδριάση του ΕΛΚ. Κάνουμε τώρα μία διακοπή γιατί η κυρία Σμιτ η αναπληρωτή, γενικό διευθυντή των εξωτερικών υποθέσεων έρχεται στι 10. Έχετε καιρό μέχρι τι 10. Ελπίζω να έχει έρθει ο πρόεδρο μα. και να προεδρεύσει όπω ήθιστε. Vielen